Το συγγνώμη κυρία Μπατζέλη, φτάσαμε επιτέλους και στη δική σας έκθεση με θέμα τις τιμές των τροφίμων στην Ευρώπη. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τους κοιόδης εισηγητές στην Επιτροπή Γεωργίας αλλά και τις τέσσερις συναρμόδιες επιτροπές της Επιτροπής, της Κομισιόν οι οποίες πραγματικά συνεργαστήκαμε για την έκδοση αυτής της έκδοσης Κύριε Επίτροπε, ήταν πάρα πολύ απλό να θέσουμε ένα ερώτημα στους καταναλωτές αν πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ για να αγοράσουν γάλα ή ένα γιαούρτι γιατί το αγοράζουν. Για το γάλα, για το γιαούρτι ή για το μπουκάλι και το κεσέ. Το ερώτημα αυτό σας το θέτω διότι στους καταναλωτές τα τελευταία χρόνια έχει περάσει έντεχνα η αντίληψη και η νοοτροπία ότι αγοράζουν ένα τρόφιμο στο οποίο μεγαλύτερη βαρύτητα έχει η ίδια η βιομηχανία που το μεταποιεί το εμπορεύεται το διακινεί παρά το ίδιο το γεωργικό προϊόν η πρώτη ύλη. πριν από δεκαπέντε χρόνια η αξία του γεωργικού προϊόντος στην τελική αξία του προς κατανάλωση συμμετείχε με 50% ενώ σήμερα μόλις με 15% οι γεωργοί οι αγρότες οι κτηνοτρόφοι είναι πλέον ανώνυμες προσωπικότητες για τους καταναλωτές. η διαπραγματευτική τους δύναμη όχι μόνο στα θέματα της διαμόρφωσης της τελικής τιμής αλλά και της διατήρησης των ποιοτικών και διατροφικών συστατικών στο τελικό προϊόν υπολείπεται του ρόλου τον οποίο έπρεπε να είχαν δεν επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε διαχωριστικές γραμμές να ταξινομήσουμε τους παραγωγικούς τομείς της αλυσίδας εφοδιασμού τον αγροτικό τον μεταποιητικό τον εμπορικό τομέα εκείνο της χονδρικής και της λιανικής πώλησης σε καλούς κακούς και άσχημους γιατί πιστεύουμε ότι δεν ζούμε σε μια κοινωνία και οικονομία με χαρακτηριστικά far west αλλά σε μια οικονομία η οποία βασίζεται σε ρυθμίσεις της εσωτερικής αγοράς της, εσωτερικής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιας αγοράς που δίνει ευκαιρίες ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας όταν λειτουργεί με διαφανή τρόπο. Εδώ λοιπόν έχουμε να αντιμετωπίσουμε δύο βασικά ζητήματα με διτό χαρακτήρα πρώτον της προσέγγισης των καταναλωτών και των παραγωγών μέσα από μια ποιοτική πολιτική στον τομέα των τροφίμων αλλά και ενίσχυσης της συνδιαμόρφωσης του τρόπου για αμεσότερη προσβασιμότητα των καταναλωτών στις παραγωγικές αγροτικές περιοχές και φορείς. δεύτερον της διασφάλισης και δεν εννοώ του καθορισμού του εισοδήματος των παραγωγών και των καταναλωτών μέσω μιας διαφανούς πολιτικής τιμών που θα περιλαμβάνει υποχρεωτικές ρυθμίσεις εποπτεία όλων των ενδιάμεσων παραγωγικών τομέων στο σύνολο της αλυσίδας εφοδιασμού. και εδώ προφανώς εννοούμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε τοπικό και εθνικό επίπεδο αλλά και τις μεγάλες επιχειρήσεις μητρικές και θυγατρικές με έδρα την ευρώπη αλλά και τους εργαζόμενους οι οποίοι πρέπει όμως να λειτουργούν με όρους διαφάνειας της εσωτερικής αγοράς και όχι εκείνο των οικονομικών παραφιάδων όπως των καρτέλ και των ολιγοπολίων. σήμερα λοιπόν μεταξύ των άλλων όπου οι πραγματικές τιμές παραγωγού παρουσιάζουν μία πτώση οι τιμές καταναλωτού φτάνουν στο πενταπλάσιο στο δεκαπλάσιο των τιμών που λαμβάνει ο παραγωγός όπου ο βαθμός συγκέντρωσης του λιανικού εμπορίου αλλά και των άλλων μεταποιητικών επιχειρήσεων τετραπλασιάζεται όπου οι δυσλειτουργίες της αγοράς ε, καταβάλλεται από τους μη υγιείς όρους ανταγωνισμού κρίνεται απολύτως απαραίτητο και σκόπιμο να υπάρχει ένας ευρωπαϊκός συντονισμένος σχεδιασμός και ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στο διατροφικό τομέα από το επίπεδο του χωραφιού μέχρι το ράφι δεν θα ήταν υπερβολή κύριε επίτροπε αν η επόμενη παρέμβαση της επιτροπής μετά τη ρύθμιση και εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος να ήταν αυτή της ρύθμισης και της εποπτείας του διατροφικού τομέα ο οποίος άλλωστε πιέζεται και από κερδοσκοπικές κινήσεις του εν λόγω τομέα. οι πολίτες έχουν την εντύπωση ότι οι αλυσίδες εφοδιασμού η μεταποίηση και το λιανικό εμπόριο είναι εκείνα που ρυθμίζουν το καλάθι της νοικοκυρά και όχι αυτή η ίδια εισοδηματική πολιτική του κράτους και της ευρωπαϊκής ένωσης. πιστεύω λοιπόν ότι ψηφίζοντας την έκθεση της επιτροπής γεωργίας και αναμένοντας τις τελικές προτάσεις της επιτροπής να αντιμετωπίσουμε διαχρονικά τα προβλήματα της λειτουργίας της αγοράς τροφίμων αγοράς η οποία μαζί με την πολιτική θα πρέπει να λειτουργεί ισομερός προς όφελος των ευρωπαίων πολιτών των ευρωπαίων αγροτών των αναπτυσσόμενων χωρών και να δημιουργεί αίσθημα ασφάλεια απέναντι στους νόμους της αγοράς και τους θεσμούς. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Θα ήθελα καταρχήν ε, να ευχαριστήσω θερμά την κυρία Μπατζελή της Επιτροπής Γεωργίας που συνέταξε αυτή την έκθεση μια κρίσιμη στιγμή για την αγροπιστιστική βιομηχανία που αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί η ύφεση οδήγησε σε μια κατακόρυφη πτώση πολλών οικονομικών κλάδων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο γεωργικός τομέας κατέρευσε, οι τιμές της αγοράς καταβαραθρώθηκαν. Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή ε, στον τομέα του κρέατος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, τομείς με προστιθέμενη αξία. Ο αγροπιστεστικός κλάδος Βέβαια θα προσπαθήσει να αυλύνει τα αποτελέσματα της κρίσης και να φτάσουν τα τρόφιμα στο καταναλωτή σε πιο προσιτές τιμές. Γι' αυτό και ο αγροπιστικός κλάδος απασχολείται ιδιαίτερα με τα θέματα της ακρίβειας και αυτό ενδιαφέρει ιδιαίτερα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μια διαρθρωτική ανάλυση δημιουργεί φόβους για εκτόξευση των αγροτικών τιμών μέσω και μακροπρόθεσμα. Βελτιώνοντας την κατάσταση στον αγροπιστικό κλάδο θα μπορέσουμε να αποφύγουμε στο μέλλον ε, μεγάλη ακρίβεια των ε, τροφίμων ή τουλάχιστον ε, μετριασμό της αύξησης αυτής. Συμμερίζουμε τις περισσότερες ανησυχίες μας, ανησυχίες ό,τι αφορά την ανάγκη βελτίωσης της γενικής λειτουργίας αυτού του κλάδου, να ενισχύσουμε τη διαφάνεια σε όλες τις φάσεις της αλυσίδας και να κατανείμουμε την προστιθέμενη αξία σε όλα τα τμήματα του κλάδου. Από πέρυσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε πολλέ πρωτοβουλίε προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργία του αγροεπιστηστικού κλάδου και μάλιστα έχουμε την ομάδα υψηλού επίπεδου για την ανταγωνιστικότητα του κλάδου ε, με πρόσφατε στρατηγικέ συστάσει. Έχουμε και μια πράσινη βιβλία για την ποιότητα των γεωργικών προϊόντων που υπευλήθη πέρυσι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην ανακοίνωση για την ακρίβεια των τροφίμων του περασμένου Δεκεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε με τη μορφή ενό φίλου πορεία διάφορε προτάσει για τη βελτίωση τη λειτουργία του αγροεπιστηστικού κλάδου στην Ευρώπη. Είναι σημαντικό να εφαρμοστεί αυτός ο δικός χάρτης και κυρίως να εφαρμοστεί να εγκαθιδρυθεί ένα ευρωπαϊκό παρατηρητήριο που θα ασχολείται με την παρατήρηση των τιμών. Θα πρέπει να παρατηρήσουμε τις ε, τιμές από την αρχή μέχρι το τέλος της αλυσίδας, ε, διευκολύνοντας την ανάλυση και, την, και εξασφαλίζοντας τη διαφάνεια. Θα πρέπει επίσης να δούμε την ευθύνη όλου του κλάδου τη αγορεπιστικής Βιομηχανία. Θα πρέπει επίσης να βελτιώσουμε τον την διαπραγματευτική ισχύ του παραγωγού που μερικές φορές γίνεται έρμος στις μεγάλες αλυσίδες. Θα πρέπει να δούμε μια πιο δίκαιη κατανομή του, του, της προστιθέμενης αξίας και μια επανισορρόπηση του διαπραγματευτικ... της διαπραγματευτικής ισχύω ε, σε όλες τις φάσεις της αγροεπιστιστικής αλυσίδας. Δεν θα πρέπει ένα τμήμα της αλυσίδας να καρπώνεται το ωφέλης βάρος ε, των παραγωγών. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε μια βιώσιμη πλατφόρμα γεωρικής παραγωγής ε, και ανταγωνιστική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να εφαρμοστεί ο δικό δικός τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πιστεύω ότι έτσι θα αντιμετωπίσουμε τι περισσότερε ανησυχίε ε, που εξέφρασε η κυρία Μπατζέλη στην έκθεσή τη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η ψηφοφορία για την έκθεση αυτή προβλέπεται να γίνει την Πέμπτη. Δίνω το λόγο τώρα στην κυρία Μπάντια Ικουτσέτ για τις καλλιτεχνικές σπουδές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η καλλιτεχνική παιδεία είναι υποχρεωτική σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές στον τρόπο με τον οποίο